διαδικασία από την ομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών, της ομάδας της αριστεράς και των ε, μη εγγεγραμμένων, έχουμε προτάσεις σχετικά με μέλη που θα οριστούν στις επιτροπές. Θα δημοσιευτεί ο κατάλογος. Αν μέχρι την ε, έγκριση των πρακτικών δεν υπάρξουν ενστάσεις, οι διορισμοί θα θεωρηθούν ε, βέβαιοι. Με βάση το άρθρο 74 του κανονισμού, ε, μαζί ε, υπέγραψα ε, τέσσερις νομικές πράξεις οι οποίες έχουν